Ε. Η Κομισιόν καλείται να πληρώσει παρακαλώ για τη φωτογραφία που θα τη βγάλουμε.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 Ready? ich bin jetzt gerade die Kamera nicht anfassen. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι έχουν παρουσιαστεί στην φωτογραφική μηχανή. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας καθυστερήσω. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1956 έλαβε χώρα σήμερα, αυτή τη μέρα, μια σημαντική επανάσταση στην Ευρώπη ήταν η εξέγερση της ε, Ουγγαρίας.